Καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας με την κυρία Μαρή Γκόγκεν Κουίν, η οποία είναι επίτροπος για την έρευνα, την καινοτομία και τις επιστήμες και τον διερθωμένο διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε την Επίτροπο που είναι σήμερα μαζί μας καθότι η συζήτηση και η συνάντησή μας προβλέπεται να διαρκέσει μία ώρα. Θα δώσουμε λοιπόν ως συνήθως για 15 λεπτά το λόγο στην Επίτροπο και μετά θα έχουν το λόγο οι επικεφαλείς αντιπροσωπιών, δηλαδή οι συντονιστές και οι συνάδελφοι που θα ζητήσουν να παρέμβουν για δύο λεπτά. Να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω με την Επίτροπο. Κάναμε υπομονή λίγα λεπτά για να προσέλθουν περισσότεροι συνάδελφοι, αλλά σίγουρα θα έρθουν εντωμεταξύ. Εντωμεταξύ μας συγχωρείτε που δεν είναι γεμάτη η αίθουσα, αλλά όσοι πιο πολύ ενδιαφέρονται για αυτό το τομέα είναι ήδη εδώ. Ε, κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Σαρτόρη, αγαπητοί βουλευτέ. Σα ευχαριστώ για την ευκαιρία να συναντηθούμε σήμερα στο πλαίσιο του διαφορμένου διαλόγου. Όπω όλοι γνωρίζουμε, η οικονομική ανάκαμψη τη Ευρώπη και η μακροπρόθεσμη ευημερία τη ε, εξαρτάται από τη δυνατότητά μα να ε, τονώσουμε την κοινοτομία με νέε ιδέε για προϊόντα, υπηρεσίε και ε, θέσει εργασία, καλύτερε ζωέ για του ανθρώπου στην Ευρώπη το 2013. Για να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση, θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέε θέσει εργασία και παραγωγικότητα σε νέο επίπεδο. Με συγχωρείτε, αλλά ενώ προσπαθώ να σα ακούσω από τα ακουστικά για να έχω καλύτερο ήχο, δεν ακούγονται αγγλικά. Στο μηδέν. Ah, eh, Κάποιο στην αίθουσα λέγει, λέει ότι δεν φτάνει η διερμηνία. Για ένα λεπτό ή διακοπή τουλάχιστον αν θέλετε να αλλάξετε θέση. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι δεν φαίνεται να έχουν πρόβλημα. Πρέπει.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 Θέλουμε να δημιουργήσουμε λοιπόν μια ανοιχτή οικονομία που να δημιουργεί καινοτομία για καινοτόμου επιχειρηματίε. Θέλουμε παραγωγικέ επενδύσει, ώστε να υπάρχει τέτοια οικονομία που να δημιουργήσουν μικρομεσαίε επιχειρήσει ευημερία. Αυτό σημαίνει ότι έρευνα και καινοτομία πρέπει να θερίζεται σε ένα δημόσιο τομέα, ο οποίο αναζητεί τρόπου για να καινοτομήσει και να επενδύσει στην καινοτομία μέσω προεμπορικών ε, ε, προεμπόρευση, ε, προμηθειών πρώτου σταδίου τη εμπόρευση. Έτσι λοιπόν η καινοτομία θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη και τι θέσει εργασία για την επιτυχία τη Ευρώπη το 2020. Αυτά βέβαια θα εξαρτηθούν από την έρευνα και την καινοτομία εφόσον είναι εύρωστε. Η κρίση έχει δείξει το εξή. Τα κράτη-μέλη που έχουν επενδύσει περισσότερο στην έρευνα και ανάπτυξη και την παιδεία έχουν αντιμετωπίσει καλύτερα τι ε, οικονομικέ αναταράξει. Γι' αυτό το Horizon 2020 θα έχει στόχο να προωθήσει την έρευνα και καινοτομία στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ο πρώτος στόχος ε, παγκοσμίως, ο πρώτος προορισμός παγκοσμίως, για να μπορέσουν ε, οι επενδύσεις να στηρίξουν τις ευρωπαϊκές πολυεθνικές και να προσελκύσουμε ξένες άμεσες επενδύσεις. Αυτό σημαίνει ότι έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη και να είμαστε ανταγωνιστικοί και στο μέλλον. Αυτό απαιτεί προστασία και ενδυνάμωση των δημόσιων προμηθειών στην έρευνα και ανάπτυξη και επιτάχυνση των πολιτικών εικόνα πρώτη ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Πρέπει να έχουμε σταθερέ μακροπρόθεσμε προοπτικέ για του επενδυτέ και του ερευνητέ παγκοσμίω, ώστε να του πείσουμε ότι το να επενδύσουν και να εργαστούν στην Ευρώπη τώρα είναι κατάλληλη επιλογή. Με ένα κατάλληλο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και το Horizon 2020 και τον κατάλληλο προπολογισμό του, μπορούμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα για τι κοινέ δεσμεύσει τη Ευρώπη να παραμείνει πρώτη στην έρευνα και την καινοτομία. Εάν δεν δώσουμε αυτό το μήνυμα, μπορεί να χάσουμε την εμπιστοσύνη που έχουν σε εμά οι επενδυτέ σε όλο τον κόσμο και να διακινδυνεύσουμε την ανάπτυξη και τι θέσει εργασία που τόσο πολύ χρειαζόμαστε. Παρά το γεγονό ότι τα ποσά που συμφωνήθηκαν το Φεβρουάριο από του ε, επικεφαλεί κρατών και κυβερνήσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτω από το επίπεδο που είχε επιθυμήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολιτικέ συμφωνίε μπορούν ακόμη να προσφέρουν ε, τόνωση στον τομέα τη ανάπτυξη και των θέσεων εργασία. Τα συμπεράσματα της Συνόδου στήριξαν τους στόχους του Horizon 2020 και εδώ παραθέτω τι έλεγαν τα συμπεράσματα, ότι η ευφυής και συνολική ανάπτυξη σημαίνει ότι θα δώσουμε προστιθέμενη αξία σε ένα τομέα που χρειάζεται δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προγράμματα που έχουν συμβάλει στην επιδίωξη των στόχων της Ευρώπης το 2020 μπορούν να συνεισφέρουν ιδιαίτερως στους στόχους της στρατηγικής αυτής με την χρηματοδότηση του Horizon 2020 και του Erasmus για όλους. Προγράμματα που μπορούν να δώσουν πραγματική ανάπτυξη σε σχέση με τα επίπεδα του 2013. Τέλος του παραθέματος. Εδώ τα συμπεράσματα δεν έχουν δώσει συγκεκριμένους αριθμούς βέβαια για το Horizon 2020, όμως η συμφωνία που επετέφθη υπονοεί έναν αριθμό γύρω στα 70 δις για τα επερχόμενα 7 χρόνια. Αυτό σημαίνει μια αύξηση περίπου 25% σε σύγκριση με τι αντίστοιχε δραστηριότητε υπό το τρέχον ε, δημοσιο... πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και αυτό βέβαια είναι χαμηλότερο από τα 80 δι ευρώ που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολύ λιγότερο από τα 100 δι ευρώ που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά θα αναλύσουμε λεπτομερώ αυτόν τον αριθμό για να δούμε πώ θα σχεδιαστεί αναλόγω το Horizon 2020. Κατά κύριο όμω λόγο, πρέπει πλήρω να σεβαστούμε το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να εκφράσει τι απόψει του σε σχέση με το ζήτημα αυτό κατά τη διάρκεια τη ε, έγκριση. Η προηγούμενη απόφαση που έλειφθη στην Ολομέλεια του Στρασβούργου έδωσε ένα ηχηρό μήνυμα μαζί με τι γενικέ κατευθυντήρε γραμμέ που στείλατε για, για τη διαχείριση της, ε, του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2014. Βεβαίω, η αβεβαιότητα δεν είναι κάτι καλό για του ε, ενδιαφερομένου και εταίρου. δημοσιονομική Ιταλικές αρχές φέτος δεν θα μπορέσουν να ξεκινήσουν καμία διαδικασία για αποβολή προτάσεων για το 2013. Και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει περικοπή 10% στι συνολικέ δημόσιε δαπάνε για την έρευνα και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση απευθεία. Δεδομένη τη σημασία τη έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη χρηματοδότησή τη για πολλά πανεπιστήμια, καθώ και ερευνητικά κέντρα σε όλη την Ήπειρο, αυτό σημαίνει ότι θα δώσουμε ένα πολύ δυνατό πλήγμα στο όλο σύστημα. Στηριζόμαστε στους βουλευτές για να, βεβαιωθούν ότι δεν θα για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα προκύψει κάτι τέτοιο. Γνωρίζω ότι οι διαθεσμικές διαπραγματεύσεις πηγαίνουν σχετικά καλά. Ήθελα εδώ να ευχαριστήσω την πρόεδρο Σαρτόρη και τους συζητητές ε, της Επιτροπής σας γι' αυτό. Στην τελευταίο τριμερή διάλογο στις 5 Μαρτίου επιτύχαμε συγκεκριμένη πρόοδο για μια σειρά από άρθρα στα πλαίσια του προγράμματο πλαισίου. Επίση, γνωρίζω ότι χρειάζεται περισσότερη εργασία για συγκεκριμένα ζητήματα, όπω σε σχέση συνεργασία με τα διαφορετικά ταμεία, πάνελ επιστημονικών και στρατηγικών ε, συνεργατών, τα, τα εργαλεία για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, την καινοτομία, τι ε, εταιρικέ σχέσει δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, και είμαι βέβαιο ότι θα καταλήξουμε σε μια ισορροπή συμφωνία για όλα αυτά τα ζητήματα. Όμω εδώ θέλω να δώσω έμφαση στο εξή. Για άλλη μια φορά σήμερα. Υπάρχει απόλυτη ανάγκη να υπάρξει χειροπιαστή απλούστευση. Η απλούστευση είναι κάτι που συμπεριλήφθη στο σχεδιασμό του Horizon 2020 και στα περιεχόμενα των συγκεκριμένων στόχων του και βεβαίω και στου κανόνε συμμετοχή και διάδοση. Πρέπει η χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής έρευνας να γίνει απλούστερη και συνεπέστερη. Έτσι, το Horizon 2020 θα μπορέσει να είναι πιο φιλικό και προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να ε, είναι ανοιχτό σε νέους συμμετέχοντες. Αυτό σημαίνει διάδοση τεχνογνωσίας που είναι απαραίτητη για την ε, καινοτομία και τον σχεδιασμό πολιτικής. Χρειάζεται ένα κοινό σύνολο κανόνων που να καλύπτει την επιλεξιμότητα, την, ε, υποβολή, τη λογοδοσία, την υποβολή εκθέσεων, τον έλεγχο και αυτό να ισχύει παντού. Χρειάζεται ένα ελάχιστο πλαίσιο ευελιξία ώστε να καταγράψουμε τι συγκεκριμένε ανάγκε συγκεκριμένων πρωτοβουλειών, όπω τα JTI. Προκειμένου να υπάρχει λιγότερο διοικητικό άχθο για του δικαιούχου και τα προγράμματα να γίνουν ελκυστικότερα, χρειάζεται μια ριζικά απλουστευμένη προσέγγιση για την ε, επιστροφή του κόστου. Αυτό βασίζεται στο ε, κατά πόσον θα γίνουν αποδεκτέ οι συνηθισμένε πρακτικέ λογοδοσία και διαχείριση των δικαιούχων με συγκεκριμένα ποσά κατά Η προσέγγιση τη Επιτροπή, ένα σχέδιο, ένα ποσοστό χρηματοδότηση και ένα κατά ποσό για το έμεσο κόστος είναι ακρογωνιαίος λήθος για την απλούστευση. Για παράδειγμα, το σύστημα 100 προς 20 χρησιμοποιήθηκε από το, για το δημοσιονομικό πλαίσιο, ε, για το πλαίσιο πρόγραμμα πλαίσιο μάλλον 7 για την έρευνα και την ανάπτυξη, κάτι που ήταν ε, πολύ ευρεώς αποδεκτό από τους ενδιαφερομένους, ιδίω τα πανεπιστήμια και τους ε, ενδιαφερομένους οργανισμούς. Η πρόταση λοιπόν αυτή θα πρέπει να στηριχθεί από τον ε, σχετικό τομέα, εάν θέλουμε να τονώσουμε την έρευνα και την καινοτομία μέσω του Horizon 2020. Οι δικαιούχοι θα κερδίσουν πολλά από την απλούστευση την, τον περιορισμό του δικαιτικού άκθους και την νομική βεβαιότητα για το κόστος που θα ζητούν να επιστραφεί και με χαμηλότερα ποσοστά σφάλματος. Τα σημεία αυτά τονίστηκαν και από το ελεγκτικό συνέδριο στη γνωμοδότησή του για του κανόνε συμμετοχή. Καταλαβαίνω ότι δεν έχετε αρχίσει ακόμα να συζητάτε το μοντέλο χρηματοδότηση του τριμερού διαλόγου σα. Είμαι όμω βέβαιη ότι οι πτυχέ αυτέ θα ληφθούν επαρκώ υπόψη όταν θα αρχίσετε τι διαπραγματεύσει σα τον επόμενο μήνα. Να σα διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει πλήρω δεσμευμένη να συνεχίσει τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να δημιουργήσουμε το δρόμο για μια πραγματική συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση και έγκαιρη έγκριση του Horizon 2020 και τη δέσμη μέτρων του. Για τι υπόλοιπε πρωτοβουλίε, με μεγάλη χαρά να σα ενημερώσω ότι οι πρωτοβουλίε για την έρευνα και την ανάπτυξη που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2012 είναι έτοιμε εγκαίρω με μία εξαίρεση. Την ανακοίνωση για την κατάσταση τη καινοτομία στην Ένωση το 2012. Αυτή θα εγκριθεί αυτή την εβδομάδα και γι' αυτό θα επανέλθουμε αργότερα. Η ανακοίνωση αυτή για την ERA e και την ε, και η ανακοίνωση για τη διεθνή συνεργασία σε έρευνα και καινοτομία θα εγκριθούν τον Ιούλιο και Σεπτέμβριο 2012 όπω προβλεπόταν και θα υλοποιηθούν αναλόγω. Οι προετοιμασίε νομοθετικών προτάσεων για τι εταιρικέ σχέσει, σχέσεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα και δημόσιο-δημόσιου τομέα έχουν ανακοινωθεί στο πρόγραμμα εργασιών μας για το 2013. αυτέ ετοιμάζονται ήδη και μάλλον θα εγκριθούν νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε προκειμένου να διευκολύνουν τι διαθεσμικέ διαπραγματεύσει και την έγκριση ε, πριν από τι ευρωεκλογέ. Και οι δύο αυτέ νομοθετικέ προτάσει έχουν ένα κοινό στόχο. Να δημιουργηθούν σχέσει συνεργασία στα πλαίσια του Horizon 2020. Σχέσει συνεργασία που θα φέρουν κοντά ευρωπαϊκά και εθνικά ευρωπαϊκούς εθνικούς φορείς με σχέσεις συνεργασίας ε, δημόσιου και δημόσιου τομέα αλλά και με, σχέ, με συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα. Παρά τις περικοπές του προπολογισμό θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των υπερχόντων πόρων, να ενισχύσουμε τις επενδύσεις και να έχουμε κρίσιμη μάζα για τις ενισχυμένες σχέσεις συνεργασίας στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας προκειμένου να πετύχει και η Ένωση της Καινοτομίας. Η διαδραστική σχέση μεταξύ των εταίρων που έχουν διαφορετικές σκοπιές θα τονώσει τον ε, αντίκτυπο του Horizon 2020 βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα του τομέα, διευκολύνοντας την ανάπτυμπόρευση νέων τεχνολογιών και νέων προϊόντων σε καθοριστικούς τομείς όπως η φαρμακολογία, η ενέργεια, οι μεταφορές, η ηλεκτρονική, η αεροπ και η βιο... βιομηχανία που βασίζεται σε βιολογικά προϊόντα. Οι σχέσεις αυτές συνεργασίας θα αποφύγουν τον κατακαιρματισμό και θα δημιουργήσουν νέες σχέσεις προκειμένου να μεταφραστεί η επιστημονική μα πρωτιά και σε βιομηχανικά πλεονεκτήματα. Και βεβαίω αυτό θα επιτρέψει οικονομική ανάπτυξη και καινοτόμε λύσει σε μεγάλα προβλήματα τη κοινωνία. Οι νέε εταιρικέ σχέσει θα πρέπει να είναι πολύ φιλόδοξε και να λειτουργούν απευθεία ε, εύρυθμα από την αρχή τη ε, ε, υλοποίησης του Horizon 2020. Οι υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται με του διάφορου ενδιαφερόμενου φορεί διάφορους για να πετύχει η προετοιμασία και θα παρουσιάσουμε το σύνολο των προτάσεων στο τέλο Ιουνίου. Οι νέε εταιρικέ σχέσεις θα λάβουν υπόψη τα διδάγματα που έχουμε από τις ισχύουσες εταιρικέ σχέσεις συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των ενδιάμεσων αξιολογήσεων, των συστάσεων των ε, διαφορών φορέων και ενδιαφερομένων και τι συνεχιζόμενε μελέτε αντικτύπου. Η χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τι μελλοντικέ σχέσει συνεργασία θα βασιστεί σε κοινέ αρχέ για την ε, σωστή διαχείριση, την διαφάνεια, τον ανοιχτό ανταγωνισμό και την αριστεία. Οι κανόνε του Horizon 2020 για τη συμμετοχή και την διάδοση θα συνεχίσουν να ισχύουν. Μπορεί να υπάρχουν συγκεκριμένε λειτουργικέ ανάγκε, οπότε να υπάρξουν και κάποιε συγκεκριμένε εξαιρέσει από αυτού του κανόνε. Αυτέ θα δικαιολογηθούν σε ελάχιστο βαθμό. Η δεύτερη επίσης έκθεση για την κατάσταση της καινοτομία στην Ένωση που θα υιοθετηθεί αυτή την εβδομάδα παρουσιάζει τις πρώτες πολιτικές προτεραιότητες και τα επιτεύγματα που ε, είχαμε το 2012 προκειμένου να δώσουμε αποτελέσματα στις 34 δεσμεύσεις για την ε, σφαιρική, την συνολική στρατηγική της καινοτομίας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ ευχαριστώ εκ μέρους όλων των συναδέλφων, την Επίτροπο. Ξεκινάμε τώρα τη συζήτησή μας με την Πιλάρ Δεκθυγιο του ΕΛΚ. Gracias, Presidenta. Bienvenida una vez más a la Comisión, Comisaria, en esta... Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας για άλλη μια φορά. Ουσιαστικά έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος της θετίας μας. Και η πιο σημαντική πτυχή η οποία μας απασχολεί είναι φυσικά το πρόγραμμα Horizon 2020. Γιατί έχει στο στόχαστρο θέματα απασχολησιμότητας, ανταγωνιστικότητας και νοτομίας. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια φάση έντονης κρίσης, η οποία πλήττει πιο πολύ κάποιες χώρες από ό,τι άλλες πλήττει ιδιαίτερως και τους ερευνητές σε όλα τα κράτη-μέλη. Ορίζοντας λοιπόν 2020 διασφαλίζει το μέλλον, μια βασική υποστήριξη σε ό,τι αφορά τις ε, δημοσιονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό ήθελα να τονίσω δύο στοιχεία τα οποία μας απασχολούν ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Εκατό δις ζήτησε το, Κοινοβούλιο, 80 δις πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόκειται για μεγάλη διαφορά. Θεωρώ παράλληλα αυτά ότι θα έπρεπε να προσπαθήσουμε στο βαθμό του δυνατού να πετύχουμε μια συμφωνία. Οι συνάδελφοι που ήταν εισηγητές από πλευράς του Κοινοβουλίου για τα θέματα αυτά διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο και θα πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο, να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να είναι συντονισμένη η προσέγγιση μας. Θα ήταν ε, πραγματικά πρόβλημα να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ε, για το θέμα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω πόσα χρήματα διατίθενται στην τελική ανάλυση. 4 δις πάνω, 4 δις κάτω, ενδεχομένω νομίζω ότι δεδομένης ε, τη σημερινή οικονομική κατάσταση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να θέσει και θέματα προτεραιότητα. Αυτό εξαρτάται και από τα ποσά που διατίθενται. Και άρα το 5% περισσότερο ή λιγότερο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πότε λοιπόν θα γνωρίζουμε τα πραγματικά ποσά, γιατί φυσικά αυτό επηρεάζει και το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Η Τερέτα Μαντουρέλ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Χαίρομαι ιδιαίτερο που, που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Και η ομάδα μου ασφαλώς ε, συμφωνεί με τις πιο πολλές σκέψεις τις οποίες παρουσιάσατε και σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα για το πρόγραμμα Horizon 2020. Αυτό ασφαλώς είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ερευνητές και τις ερευνήτριές μας το πρόγραμμα αυτό. Να ξεκινήσω τονίζοντας τα θετικά στοιχεία τα οποία αναφέρετε και εσείς άλλωστε. Είμαστε ιδιαίτερως ικανοποιημένοι σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για τον ορίζοντα 2020, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Τα πιο σημαντικά στοιχεία του διτακτικού έχουν αποφασιστεί και στα υπόλοιπα θέματα φαίνεται ότι σημειώνεται πρόοδος. Δεν πρόκειται να επισέλθω σε λεπτομέρειε, τα, κάνατε, τα αναφέρατε εσεί άλλωστε. Στι 8 Μαρτίου ήταν Διεθνή ημέρα, Παγκόσμια ημέρα τη γυναίκα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να τονίσω ότι θα έπρεπε να σημειωθεί πρόοδος και σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων και σε ό,τι αφορά και την πρόσβαση στις δημοσιεύσεις. Αυτό φυσικά σχετίζεται και με τα θέματα ανταγωνιστικότητας. Η γυναίκα θα πρέπει να συμμετέχει πιο έντονα. Γιατί στον τομέα αυτό μπορεί να αναδειχθεί και η γυναικεία δημιουργικότητα και αυτό με τη σειρά του μπορεί να ε, τονώσει και την οικονομία. Θα ήταν απαραίτητο επίσης η διαδικασία καινοτομία να υποστηριχθεί σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι άλλο τώρα που θα ήθελα να αναφέρω. Θίξατε κι εσείς το θέμα αυτό. Το έθιξε και η συνάδελφος. Είναι ένα θέμα που απασχολεί και την ομάδα μας. Μιλάω για τις αμφιβολίες που επικρατούν για τη γραμμή του προπολογισμού 1α. Πρόκειται για κάτι το οποίο αντιτίθεται στις ε, απόψεις του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά και με θέματα και στόχους που έχουν τεθεί για την ανταγωνιστικότητα και την ε, ανάπτυξη. Όλοι όσοι ασχολούνται με το πρόγραμμα από όλες τις ομάδες θέλουν πραγματικά να προασπιστούν ε, έναν ελάχιστο προϋπολογισμό για το πρόγραμμα αυτό από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ως εισηγήτρια του προγράμματος Ορίζοντας 2020 πρέπει να σας πω ότι και το Κοινοβούλιο ασφαλώς στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας θα μπορούσε να διοργανώσει προγράμματα σε διασυνοριακό επίπεδο, το οποίο θα ωφελούσε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε διάφορες περιπτώσεις ακούστηκαν θέματα ε, αδιαφάνεια σε ό,τι αφορά τα TTIs. Τέλος, ε, πρέπει να ρωτηθούμε πώς μπορούμε να ε, προωθήσουμε τα προγράμματα αριστείας. Ε. Πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την πρόσβαση στον ορίζοντα 2020. Συμφωνείτε ότι θα πρέπει να εγγυηθούμε θέματα διαφάνεια σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα προγράμματα αυτά και στα GTIs μπορείτε να μας ε, παρουσιάσετε τα αποτελέσματα της μελέτης αντικτύπου για τα GTI, η οποία η μελέτη έγινε προσφάτως για να βρούμε νέες λύσεις για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τζόρντιν για δύο λεπτά. Τώρα έχει το λόγο λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο κατηγορίες ερωτήσεων θα ήθελα να σας απευθύνω. Η πρώτη κατηγορία έχει να κάνει με την προώθηση της αριστείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζω έντονα το στόχο αυτό, όπως και όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άλλωστε. Ένα, πρόγραμμα, ένα τμήμα του προγράμματος έχει διαμορφωθεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να προωθηθεί ακριβώς ε, ο σκοπός αυτός. Ένα δισεκατομμύριο θα χρειαζόμασταν. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι σαφή η τοποθέτησή σας για τον προϋπολογισμό. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο συμφωνείτε με τη δική μας άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ποιες αρχές υποστηρίζετε κατά την κατανομή πιο πολλούς ε, στόχους με λιγότερα χρήματα ή λιγότερες πρωτοβουλίες με τα λιγότερα χρήματα. Αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερη κατηγορία ερωτήσεων τώρα σε ό,τι αφορά τα flagships. Τα υποστηρίζω φυσικά ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά την σύνδεση μεταξύ γνώσης και τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερως και θα πρέπει να το προωθήσουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προγράμματα τα οποία έχουν υποστηριχθεί είναι από 15 κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μου πείτε πώς θα φροντίσετε ε, ότι θα αναπτυχθεί όλο το ευρωπαϊκό δυναμικό. Και θα μείνουν ανοιχτέ οι πρωτοβουλίε αυτέ. Ευχαριστώ πολύ. Η Μαρία Καρβαλιό. Ευχαριστώ, κυρία Σαρτόρη, επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας να επικεντρωθώ στις διαπραγματεύσεις για το Horizon 2020. Εναρκτήρια συνάντηση για τον τριμερή διάλογο έγινε ε, τα τρία θεσμικά όργανα εξέφρασαν την δέσμευσή τους και την διάθεση να επιτύχουν συμφωνία σε βασικούς τομείς. Έχουμε επιτύχει κάποια πρόοδο, ιδίως όπως ανέφερε και η Επίτροπος Γκίγκαν. Ο τελευταίος τριμερής διάλογος ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικός και επιτύχαμε πρόοδο σε διάφορα θέματα. Πολλά ζητήματα βέβαια, η συζήτηση πρέπει ακόμη να γίνει. Αναφέρατε και εσεί σημαντικά θέματα που ακόμη δεν έχουν επιληθεί επίτροπε, όμως ήθελα να προσθέσω και εγώ κάτι. Κάτι πολύ σημαντικό και για το Ευρωκοινοβούλιο και όπως το είπε και η κυρία Τζόρνταν, είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή η δική μου συγκεκριμένα έκθεση, αυτή που ετοιμάζω, μιλά για συγκεκριμένες δράσεις όπως ε, την, ε, ε, το σχηματισμό ομάδων, ή σχέσεις με δύο τουλάχιστον φορείς για την πρόθεση πρωτοβουλειών που για μας είναι πολύ σημαντικές. Επίσης, ζητούμε συγκεκριμένη δημοσιονομική γραμμή για τις δράσεις αυτές και τη στήριξή σας. Στήριξη για την στρατηγική που προτείνουμε, συμπεριλαμβάνοντας αυτές τις συγκεκριμένες ε, δωρεές, αυτές τις συγκεκριμένες, αυτά τα συγκεκριμένα ποσά στήριξης. Το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Να σας ρωτήσω για αυτό το ποσό που αναφέρατε για το ορίζον 2020 βεβαίως και υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και επί τη βάση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου επίσης ε, υπάρχει και μια φράση που λέει ότι ε, το 2020 θα πρέπει με σχέση με το επίπεδο 2013 να είναι διαφορετικό, να είναι αναπτυξιακό. Οπότε αν λάβετε υπόψη ε, το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και αυτά τα οποία εκεί καλύπτονται τουλάχιστον όπως εγώ το υπολογίζω τελικά. Πάμε πάνω από τα 70 εκατομμύρια, τουλάχιστον όπως το υπολογίζω εγώ. Άρα και εμείς ελπίζουμε να είναι το ποσό ανώτερο. Και επίσης θα θέλαμε να μας δώσετε κάποια ελπίδα από κάποιους υπολογισμούς και να επιβεβαιώσετε ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Ευχαριστούμε. Έλερ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, πρόεδρο Σαρτόρη γιατί παρά το γεγονός ότι ασκήθηκε έντονη πίεση υποστηρίζει τις κοινέ θέσει του Κοινοβουλίου και αυτό το λέω επειδή οι έως τώρα συζητήσει έγιναν με πολιτική και προσωπική υποστήριξη της Επιτρόπου. Και τώρα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι όπου δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να παίξει τον δίκαιο διαμεσολαβητή μεταξύ ημών και του Συμβουλίου και στο μέλλον. Να δώσω ένα παράδειγμα. Στις τεχνικές ε, αν κάνουμε μία πρόταση με την οποία θα συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο, και θα πρέπει να ε, οριστεί για παράδειγμα ότι θα πρέπει να διατίθενται στους υποψηφίους ε, τα ε, σχετικά έγγραφα και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τεχνική συνάντηση αναφέρει ότι αυτό είναι η κόκκινη γραμμή, εμείς τι θα κάνουμε, τρεις δυνατότητες, ή θα καταγγείλουμε στο δικαστήριο, είτε θα πούμε ότι θα πρέπει να το επιλύσει αυτό το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα, ανεπιμείνει ότι το θέμα αυτό είναι ανεπίλητο από πλευρά του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να ζητήσει ε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις. Ελπίζω να μείνουμε σε αυτό το θετικό κλίμα, αλλά θα ήθελα να πω ότι ως όροι ε, για τη συζήτηση. Έχουν τεθεί κάποιες γραπτές ερωτήσεις, οι οποίες ακόμα δεν έχουν απαντηθεί, αλλά είναι πολύ απαραίτητο να απαντηθούν για να ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Και πώς θα προχωρήσουμε. Ένα τελευταίο θέμα που με απασχολεί σε ό,τι αφορά και αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Ε, το θέμα του ορίζοντα 2020. Δεν έχουμε όμως τα αριθμητικά στοιχεία για το 1α. Και έτσι έχουμε μια κατάσταση όπου προγράμματα όπως το GMS για παράδειγμα είναι πολύ υποχρηματοδοτημένα. Έχουν λάβει πολύ περιορισμένα κονδύλια και το θέμα λοιπόν είναι τι θα γίνει στο μέλλον. Ε. Όπως το GMS για παράδειγμα θα μπορούσαν να βγουν από το πρόγραμμα του 2020. Αυτό καταδεικνύει πόσο προβληματική είναι η κατάσταση όταν διαπιστώνουμε ότι είναι πραγματικά πολύ περιορισμένη η χρηματοδότηση για κάποια τέτοια προγράμματα. Άρα, Επίτροπε, σας παρακαλώ, μην μιλήσετε μόνο για θέματα προπολογισμού, αλλά ε, μιλήστε μας και για το βασικό θέμα, το βασικό πρόβλημα των ε, συνδεδεόμενων, αν θέλετε, τέτοιων ζητημάτων στο 1α. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλάς. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ που ήρθατε δύο παρατηρήσεις και τρεις ερωτήσεις. Στην ομιλία σας αναφέρατε ότι πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε για να εξακολουθήσει η Ευρώπη να παραμένει πρώτη στο R&D. Ποιος σας είπε ότι η Ευρώπη είναι πρώτη στο R&D. Καμία μελέτη διεθνούς οργανισμού, καμία μελέτη εταιριών, καμία από τις παραμέτρους δεν δείχνει ότι έχουμε την πρώτη θέση διεθνώς. Επομένως, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε την έκθεση για την κατάσταση της έρευνας και τεχνολογίας στην Ευρώπη που πρόκειται να παρουσιαστεί. Η κυρία Τζόρνταν έκανε αναφορά για διασυνοριακές ε, συνεργασίες ερευνητικού περιεχομένου. Είχαμε την ευκαιρία στο Στρασβούργο να ακούσουμε τον πρόεδρο του Ισραήλ, τον κύριο Σίμον Πέρες, να μας λέει ένα όνειρο όπου η τεχνολογική και επιστημονική υπεροχή του Ισραήλ συν την άθρηση διεθνών εταιριών και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να δώσει ειρήνη και ανάπτυξη στην περιοχή της Παλαιστίνης. Φαντάζομαι ότι ένα τέτοιο μοντέλο θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να το σκεφτεί και για τον εαυτό της. Σχετικό με αυτό, επομένως, είναι και το ζήτημα της, αλληλεσύν, της σύνδεσης των διαρθρωτικών ταμείων με τους γενικούς, με, τις, με τους τέσσερις πυλώνες του ορίζοντα, έτσι ώστε χρήματα τα οποία στο παρελθόν σπαταλήθηκαν να υπαχθούν στην γενική πολιτική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο θεματικά όσο και ως προς την επίτευξη της αριστείας που θα μπορούσε να βοηθήσει τις χώρες που υπολείπονται. Θέλω να σας ευχαριστήσω επίσης γιατί για πρώτη φορά ακούω να αναγνωρίζετε ότι δεν υπάρχει διαφορά Βορρανότου αλλά υπάρχει διαφορά μεταξύ των χωρών που κατάφεραν να πλησιάσουν τους στόχους της Λισαβόνας και εκείνων που απέτυχαν. Έτσι λοιπόν επιβεβαιώνεται ότι ένας από τους λόγους της οικονομικής κρίσης της Ευρώπης είναι η υποχρηματοδότηση της έρευνας και όχι το ανάποδο, ότι δηλαδή ότι η κρίση υποχρηματοδοτεί την έρευνα. Ευχαριστώ πολύ. σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, καλωσορίσω και εγώ την Επιτροπή Queen στην Επιτροπή μας. Συμφωνώ απόλυτα με τα θέματα απλοποίησης που αναφέρεται. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η απλούστευση. Κοιτώντας και την σύνδεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τα κέντρα αριστείας. Εδώ η απλούστευση, simplicity, είναι πάρα πολύ σημαντική πραγματικά. Ανακύπτει και το ερώτημα ασφαλώς του κατά πόσον θέλουμε και πώς θέλουμε να εμπορευτούμε την τεχνογνωσία μας εκτός Ευρώπης. Έχουμε μία ανταγωνιστικότητα στο εσωτερικό της Ευρώπης, στο εσωτερικό της Ευρώπης, αλλά αυτό μήπως αποδυναμώνει την Ευρώπη στο εξωτερικό. Οι τρίτες χώρες δεν μας περιμένουν εκεί, είναι η Βραζιλία. Και γι' αυτό λοιπόν έχω βασικά την εξή ερώτηση να θέσω. Πώς θα μπορούσαμε να αποδυναμώσουμε τον εσωτερικό ανταγωνισμό και να ενισχύσουμε τις συνδέσεις που υπάρχουν και πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελα να ενισχύσει την δικτύωση προκειμένου να προωθήσει και την εμπορία των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κ. Λαντ, ευχαριστώ Πρόεδρε Επίτροπε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο γιατί πολλοί συνάδελφοι το έθεσαν. Το θέμα λοιπόν είναι ο προπολογισμό. Δεν θα σα προκαλέσει έκπληξη. Ε, αναφέρεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου ότι ορίζοντα 2020 και το Εράσμου ε, θα πρέπει να κοιτάξουμε την κατάσταση του 2013. Θα ήθελα να ξέρω τι εννοεί το Συμβούλιο όταν μιλάει για ανάπτυξη. Ένα ευρώ, ένα εκατομμύριο, ένα δισεκατομμύριο και κατά δεύτερο χρειαζόμαστε τα στοιχεία του 2013 για να έχουμε μια συγκρισιμότητα. Να ξέρουμε ότι αυτά είναι τα στοιχεία για το 2013 και θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε επί 7, για παράδειγμα. Να ξέρουμε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Ευχαριστώ. Λέει σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Επιτροπή που ήρθατε να μας δείτε. Θέλω να υπονθυμίσω κάτι το οποίο καμιά φορά το ξεχνούμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε την έκθεση αυτή. Την έκθεση αυτή που αφορά κάποιες περιφέρειες, κάποιες περιοχές που ήταν βιομηχανικές. Και αυτό είναι σημαντικό διότι εκεί όταν κλείνουν οι βιομηχανίες τότε γίνονται περιοχές αστικές και όχι ε, άλλης ε, οικονομικής δραστηριότητα. Ή μπορεί να έχουμε επίσης και περιοχές που ε, γίνονται περιοχές ανάπτυξης πράσινης οικονομίας. Επομένως, έτσι μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το φαινόμενο και μπορούμε να αντιλήσουμε χρήματα από κάποια αντίστοιχα ταμεία γιατί δεν θα πρέπει να προσέχουμε μόνο τη βιομηχανία. Θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι αυτές οι περιοχές για τις οποίες μιλώ δεν θα ξαναγίνουν βιομηχανικές περιοχές. Μην το ξεχνούμε. Θα γίνουν κάτι άλλο. Θα αναπτυχθεί και κάποια άλλη δραστηριότητα. Επομένως, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να μην χαθούν θέσεις απασχόλησης με αυτόν τον τρόπο, να προσέξουμε την ε, ανάπτυξη και αυτές να τις κάνουμε ειδικέ ε, ζώνες προστασίας, ζώνες ελευθερού εμπορίου, που έχουν χαθεί πολλές τέτοιες. Και όμως θα πρέπει να προσέξουμε πολύ περισσότερο από ό,τι προηγουμένως. Ας πούμε η πετροχημική βιομηχανία και αυτή έχει χτυπηθεί και άρα θα πρέπει και εδώ να δώσουμε βάρος, να δώσουμε έμφαση στην έρευνα. Φόρντ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Πέρασε τώρα η γιορτή του Αγίου Πατρικού, όπως εγώ σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και έχω τρεις ερωτήσεις μιλούμε για 25% αύξηση όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Τότε το 25% πώς κατέληξε να γίνει 10% μείωση σε αυτά τα οποία ε, θα, θα λάβουν τα πανεπιστήμια. Όταν με ρωτάνε πώς θα τους ε, απαντήσω, εσείς μπορείτε να μου δώσετε μια απλή απάντηση. Επίσης γιατί την ανάπτυξη πάλι. Εάν έχουμε λιγότερους κανόνες σε σχέση με τη λογιστική, τότε θα υπάρχουν και λιγότερες παραβάσεις. Γιατί έχουμε βεβαίω ε, ε, αυτού που κάνουν τους ελέγχους, τους λογιστές και όλους αυτούς, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η απορρόφηση γίνεται πιο παραγωγικά. Άρα, πώς θα έχουμε αξιοποιήσει καλύτερη, γιατί έχουν πάρα πολλούς οργανισμούς οι οποίοι ε, έχουν μια, μια εύρεθμη λειτουργία και θα να συνεχίσουν να την έχουν. Επίσης, όσον αφορά το πώς έχουν κατανεμηθεί τα ε, κονδύλια του προϋπολογισμού για τη δική μας επιτροπή, βλέπουμε ότι έχουμε μείωση των ε, κονδυλίων που αφορούν την υγεία παρά το, τις τρομές εξελίξεις στο δημογραφικό. Μειώθηκε επίσης ε, η προκοδότηση για την διατροφική ασφάλεια ενώ έχουμε ε, όλο αυτό τον προβληματισμό και την ανησυχία για το τι γίνεται στην Ευρώπη για τα τρόφιμα. Οπότε μπορείτε να, να μας τα πείτε οθονομονικά θυσιαστούμε, τι γίνεται το 25%, τι γίνεται με την απλούστευση στη, στη λογιστική που δεν οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα και επίσης τι γίνεται όσον αφορά την κατανομή ή ανακατανομή των κονδυλίων του προπολογισμού. Η ανακατανομη των κωδικων του προπολογισμου η κυρια γκροστε θα έχει την τελευταία παρέμβαση, λέει ο Πρόεδρο, και μετά δώσω το λόγο στην Επίτροπο. Σα ευχαριστώ. Δύο γρήγορε ερωτησούλε. Πρώτα-πρώτα, θεωρείτε, κύριε Επίτροπε, ότι το πρόγραμμα Horizon 2020 αρκεί καλύπτει τις ανάγκες των ΜΜΕ στην Ευρώπη. Και από την άλλη μεριά ε, μιλούμε για την ε, καινοτομία, αλλά έχουμε αυτή την εκροή ε, εγκεφάλων. Πώς όλα αυτά, κάθε Πώς, πώς, πώς το βλέπετε αυτό το φαινόμενο. Θα πρέπει και τους ερευνητές μας να τους κρατήσουμε και θα πρέπει επομένως να τους πλαισιώσουμε σωστά και για αυτόν τον τρόπο να μην ε, οδηγηθούμε σε κάποιο, σε, σε κάποιο χάσμα όσον αφορά τις αμοιβέ που δίνουν κάποιες τρίτες χώρες σε αυτούς. Τι θα λέγατε. Grazie alla collega Grostet. Bene, abbiamo ε, terminato i nostri interventi. Ευχαριστούμε κύριε Κωστέ. Τελείωσαν τώρα οι παρεμβάσει και τώρα κυρία Επίτροπε, ε, νομίζω ότι το πόσο έγινε, πόσε ερωτήσει που ευλήθησαν και πόσο εύστοχε είναι δείχνουν το ενδιαφέρον μα. Οπότε σα δώσουμε ευθύ αμέσω το λόγο για τα συμπεράσματά σα. Επίτροπε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρε Σαρτόρη, πρώτα-πρώτα θα ήθελα να εκφράσω ευχαριστήσει μου προ όλου ε, οι οποίοι έλαβαν το λόγο ναι, επίση σα ευχαριστώ για το, πόσο, πόσο με υποστηρίζετε εμένα και κυρίω ε, το πακέτο ε, το, σε σχέση με τον ορίζοντα 2020 και πρέπει τελικά να γίνει σωστή πρικοδότηση για να μπορέσουμε έτσι να καλύψουμε όλες τις πλευρές του προγράμματος. Τώρα, ε, όλα αυτά τα οποία είπατε ε, όντως καταδεικνύουν το πόσο είναι κλειδί για την ανάπτυξη του Horizon 2020 και επίσης ένα αυτό το οποίο είπατε ισχύει ότι θα πρέπει να γίνει η σωστή εφαρμογή και εκτέλεσή του. Και θα ήθελα βεβαίως να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τον τρόπο με τον οποίο ο τριμερής διάλογος έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι είναι ουσιαστική εκεί η συζήτηση και ελπίζω οι υπηρεσίες που με εκπροσωπούν εκεί ε, και έτσι ε, ελπίζω ότι σας βοήθησαν έτσι όπως προχωρούμε ή στην επεξεργασία των προτάσεων τώρα θα ήθελα να συνεχίσω και να απαντήσω όσο γίνεται περισσότερες από τις ερωτήσεις και συγγνώμη κυρία Πρόεδρε εάν δεν καλύψω όλες τις ερωτήσεις αλλά αν παραλείψω κάποια ερώτηση θα απαντήσω εγγράφος. Πρώτα πρώτα να σας πω για κάτι το οποίο είπατε σε σχέση με τα δύο φύλλα. Βεβαίως ο στόχος είναι να έχουμε 50% συμμετοχή των γυναικών στις ομάδες των συμβούλων, των εμπειρογνωμόνων, στα πάνελ της, της αξιολόγησης, ε, οπότε το θέμα της όλες των φίλων θα ληφθεί υπόψη σοβαρά όταν μελετούμε τα θέματα προς έρευνα, ας πούμε σε κάποιους τομείς όπως το περιβάλλον, η υγεία κλπ. Και εγώ δεσμεύτηκα σε σχέση με αυτό ευθύ εξ αρχής Ήταν ένα από τα θέματα τα οποία μου είπατε τον Ιανουάριο του 2010 και με τους γενικούς διευθυντές τα είπαμε για να βρούμε μια σφαιρική πολιτική για όλα αυτά τα θέματα. Τώρα πάμε από το ένα στο άλλο μοιραία. Έχουμε όλες αυτές τις μέρες αξιολόγησης που είναι πάρα πολύ σημαντικές και όσον αφορά τα JTI σημαντικό για όλους μας σε σχέση δε με κάτι το οποίο είπε μια σειρά βουλευτών θα πρέπει να υπάρχει εδώ ανοιχτό χαρακτήρας να υπάρχει διαφάνεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε 100% και μάθαμε το μαθημά μας από το πρόγραμμα πλαίσιο υπαριθμών 7, να γίνει εναρμόνιση των κανόνων, ε, χρειαζόμαστε από τη βιομηχανία ξεκαθαρή δέσμευση και επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει πιο ανοιχτή διακυβέρνηση. Πήραμε το μάθημά μας, πήραμε το μήνυμα και ε, ο καθαρός ουρανός είναι ένα κλασικό παράδειγμα από αυτά που διακρίνεται από ανοιχτό χαρακτήρα. Έχουμε πάνω από 550 οποίοι εκεί συμμετέχουν. Και αυτό αποδεικνύει ότι το JTI έχει ανοιχτό χαρακτήρα. Γίνεται συνεργασία στην ε, έρευνα ε, για αυτούς τους πάνω από 550 συμμετέχοντες. 50% των επιλέξιμων είναι νέοι στο πρόγραμμα πλαίσιο. Πρόκειται για κάτι ε, που όλοι όλοι το έχουν ε, ξεκάθαρο στο μυαλό τους. θα πρέπει να έχει το Να φαίνεται τον έχει και χρειαζόμαστε και νέους συμμετέχοντες οι οποίοι έρχονται. Έχουμε δε αυτό το 40% των ΜΜΕ που έχουν μπει στο πρόγραμμα Καθρό ουρανός και συμμετέχουμε και με προτάσεις. Τώρα, άλλες ερωτήσεις που έχουν τεθεί, αυτά τα μοντέλα, τα πρότυπα χρηματοδότησης, διάφοροι από εσά είπαν κατά πόσον έχω κάποια στοιχεία στη διάθεσή μου. Ναι, στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, όπως ξέρετε, ε, τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα και με την Κομισιόν προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε αυτά τα οποία είπε το Συμβούλιο και γι' αυτό είπαμε ότι πάμε στα 70 δις ε, πάνω κάτω. Όμως αυτό είναι κάτι το οποίο το, υποθέτουμε. Θα πρέπει στον τριμερή διάλογο να συζητηθεί με Συμβούλιο και Κοινοβούλιο και βέβαια είναι σημαντικό να κατανοήσουμε το ότι κάθε δις μείωσης τι σημαίνει για το ορίζον 2020. Μια που ανέκαθεν λέγαμε ότι έχουμε τα 76-74 τέλο πάντων δηλαδή θα είναι το ελάχιστο της χρηματοδότησης που χρειάζεται εάν επιθυμούμε να μείνουμε στα επίπεδα της χρηματοδότησης του 2013 όπως ρώτησε η κυρία Καρβάλιο και άλλοι. Άρα, κοιτάξτε τι γίνεται με κάθε δις. Θα σου πω κάποια παραδείγματα και έτσι θα καταλάβετε το, το, το, την τεράστια σημασία όλων αυτών. Ας πούμε έχουμε 4.000 μνημείου που δεν θα λάβουν χρήματα για και καινοτομίε. Ή επίση σημαίνει ότι 600 άριστοι ερευνητέ και το επιτελείο του δεν πρόκειται να λάβουν τα χρήματα τα οποία χρειάζονται, ούτω ώστε να συμβάλλουν στο να έχουμε ευημερία στο μέλλον. Ή 2.500 ε, υποτροφίε στα πλαίσια του Μαρή Κιουρί δεν θα πάρουν χρήματα, δεν θα χρηματοδοτηθούν. Οπότε να δούμε αν θα μπορούσαμε να αποδημιώσουμε 10 δι ε, ω δάνεια σε ΜΜΕ και μεσαίο μέγεθος επιχειρήσει. Να, κοιτάξτε, ε, αυτό ήταν ένα δείγματάκι από τα αποτελέσματα που θα επιφέρει η μείωση του προπολογισμό. Και, όπω γνωρίζετε, έχουμε μια πάρα πολύ δυναμική πολιτική όσον αφορά την ανοιχτή πρόσβαση και τα συζητήσαμε εδώ και άλλη φορά, να μην τα ξαναπούμε. Σα ξαναλέω, οι δέσμευσή μα είναι σαφεί. Νομίζουμε ότι καλά τα πάμε και ακριβώ αυτή είναι η κατεύθυνση που έχουν λάβει όλοι στον κόσμο. Τώρα κάτι άλλο που στην εισήγησή μου όσον αφορά το ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα είναι ελκυστική προ του ερευνητέ και προ όλου του ε, επιστήμονε και να δούμε με τι κριτήρια θα προχωρήσουμε τόσο ώστε να ισχύσει κάτι τέτοιο. Για ε, κοιτάξτε, τι επενδύσει γίνονται παντού. Τι κάνουν οι ανταγωνιστέ μα, τι κάνουν, κυρίω προ Ανατολά. Τι γίνεται στην Κίνα, στη Σιγκαπούρη, στη Νότια Κορέα, τη Ρωσία. όλε αυτέ οι χώρε έχουν επισημάνει ακριβώ όπω και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η καινοτομία και η έρευνα είναι κάτι που να πάρει η οικονομία. Και επομένω οι επενδύσει σε αυτού του τομεί είναι τρομερέ. Γι' αυτό και σα λέω είναι σημαντικό η Ευρώπη να συνεχίσει και να αυξάνει τις ε, επενδύσεις τη, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε πρωτοπόροι. Έχουμε τους καλύτερους εδώ στην Ευρώπη. Έχουμε την καλύτερη έρευνα. Όμω, δεν μπορέσαμε αυτά όλα να τα μετασχηματίσουμε στην καινοτομία που θα φέρει ανάπτυξη στην οικονομία μας. Και θα πρέπει αυτό να είναι ξεκάθαρο στο ε, πλαίσιο του, του, του 2020 να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση γιατί οι ανταγωνιστές ήρθαν εδώ, δεν είναι πια εκεί πέρα μακριά. Μας ανταγωνίζονται στη συνέχεια. Απλούστευση. Από την πρώτη μέρα που ήρθε εδώ, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2010, ε, όλες οι πτέρυγες του Κοινοβουλίου μου λέγανε ότι για το πρόγραμμα πλαίσιο αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να δούμε τι θα γίνει με την γραφειοκρατία, τι θα γίνει με την κατάτμιση, τι θα γίνει με, όλα αυτά τα έντυπα, σε αιτήσει, ε, όλα αυτά πρέπει να κάνουν οι ερευνητέ, οι επιστήμονες, οι επιχειρήσεις και επομένω. συνεχώς με όλους τους εμπλεκομένους ε, συνοούμεθα και όλοι αυτό λέγανε. Πάρα πολύ, ήταν περίπου τα πράγματα, δεν φεύγανε από το πρόγραμμα πλαίσιο. Και τα πανεπιστήμια και ερευνητέ φύγαν, το άφησαν πρόγραμμα πλαίσιο και πήγαν να βρουν εθνικά κονδύλια. Τώρα επομένω τα προστέψαμε, θέλουν να επανέλθουν, αλλά ακριβώ με αυτή την προπόθεση. Αυτό το έλεγε κάθε χρόνο, εδώ και 10 χρόνια το Ελληνικό Συνέδριο, ότι θα πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία. Και ένα βασικό τρόπο να γίνει κάτι τέτοιο είναι να απλουστευτεί το πρόγραμμα. Οπότε αν υπήρχε ένα μόνο πράγμα που θα μπορούσαμε να πετύχουμε το Horizon 2000 ήταν αυτό. Να ήταν η απλούστευση και νομίζω ότι έτσι θα πετύχαινε η αποστολή μας. Και σχετικά με αυτό να ευχαριστήσω εσάς, αυτή την Επιτροπή, γιατί συνεχώς, συνεχώς με εξωθήσατε ούτω ώστε να ε, εισαγάγω όλο ένα και περισσότερη απλούστευση Γι' αυτό σας λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας στο παρελθόν και αυτή που συνεχίζει να μου δίνετε. Μου λέει η κυρία Στοτή πρέπει να κλείσω. Ελπίζω ότι κάλυψα τους περισσότερους και για τους υπόλοιπους να είστε σίγουροι ότι σε αμέσως επόμενες μέρες θα σας απαντήσω εγγράφως. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Επίτροπε, για την προσέλευσή σας και για τις απαντήσεις και για την προθυμία σας. Σε τρία λεπτάκια θα ξεκινήσουμε την διαδικασία της ψηφοφορίας. Παρακαλώ να είσαστε έτοιμοι για να χαιρετήσουμε την Επίτροπο και να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες, όχι μόνο γιατί είναι μπόλικες, αλλά γιατί είναι και μακροσκελής οι κατάλογοι. Πρώτα απ' όλα δοκιμάζουμε τις κάρτες, για να δούμε αν λειτουργούν οι κάρτες, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Πάστα. Η δοκιμή με τις κάρτες πέτυχε. Μια πρώτη πληροφορία. Στο σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης που αφορά το κοινοτικό νομικό πλαίσιο για την κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής γίνει στις 24 Απριλίου. Τότε θα ψηφιστεί, διότι εντωμεταξύ θέλουμε μια συνεννόηση να κάνουμε μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τότε θα το ψηφίσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν τις ψηφοφορίες με την έκθεση Μπέλετ. Συμβιβαστική των πολιτικών ομάδων ΕΛΚ, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Πράσινη, Άλντε, ε, συντηρήθηκε και μεταρρυθμιστές Γκουε τα λοιπά ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Η ΕΛΚ είναι κατά δύο υπεράριθμοι. Πέρας της πληροφορίας εγκρίνεται 45 υπέρ 6 κατά συγχαρητήρια. Νομοθετική πρόταση τώρα, νομοθετικό ψήφισμα μάλλον, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 43 υπέρ, 5 κατά, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Παρακαλώ κύριο Τούρμε. Δεν είχα προλάβει την κάρτα μου να βάλω, οπότε να προσθέσετε μια ψήφο και από μένα για την τελική ψηφοφορία. Ευχαριστούμε. Perfetto. Allora andiamo a votare la relazione. Και τώρα ψηφίζουμε την έκθεση Royal. Η πρώτη τροπολογία αποσύρεται. Ένα α, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ένα μπι, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για το 1B. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένα μπι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 18 υπέρ, 31 κατά. Απορρίπτεται. Με δύο αποχές. 78 υπέρ, κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. NV1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 82 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Μετά το πρώτο τμήμα, εφόσον εγκρίνεται, μπορούμε να περάσουμε απευθείας στη συμβαστική 2. Απευθείας στη συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 103. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 109 υπέρ, σε δύο τμήματα, με συγχωρείτε. 109 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 115 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ κατά αποχές 130 130 με συγχωρείτε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. 148 υπέρ κατά απόχέ. απορρίπτεται. 324 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 448 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 478 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 134 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε την 158, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 22 υπέρ, 30 κατά. Απορρίπτεται. 160. 160 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 162 υπέρ, κατά. Εκατόν εξήντα δύο. 162 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 164 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 165 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 166 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6 υπέρ, όχι, όχι, με συγχωρείτε. Έχουμε και την 337. 337 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 173. 173 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 191 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 194 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 201 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 202 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 217 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχο, έλεγχο για το 152. Votazione Χιούζα. Πέρα τη πληροφορία. 45 υπέρ 10 κατά. Εγκρίνεται. Ρέτζι 4. Πρώτο τμήμα. Σωστά. Να. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 222. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 221 με προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 223 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 υπέρ. Έλεγχο για τι πράγμα. Α, με συγχωρείτε. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. Καμιά φορά θέλετε να ελέγξουμε για την 11. Η 11 εγκρίθηκε. Δικό μου το λάθος. Μπέρδεψα τη γλώσσα μου. Για τα πρακτικά λοιπόν η τροπολογία 11 εγκρίθηκε, 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 243 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 327 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 274 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 286 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 305 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 287 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 303 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 300 151 μάλλον. 151 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 306 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Από κοινού 307 και 308 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτονται αλλά ας ελέγξουμε παρακαλώ. «307-308» πέρας σωστά αμφέβαλα, 27-26, άρα εγκρίνεται. 27 υπέρ, 26 κατά. 309 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 310 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. «325 με προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 330 και 331 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 330 έλεγχο για τα 330-31. Ωραία, έλεγχος. 330-331. Πέρας. 31 προς 24. Εγκρίνεται. 332. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πέρας. 33 προς 25 εγκρίνεται. 333 υπέρ, κατά, αποχές, ίδια διαφορά με πριν, εγκρίνεται. 334 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έλεγχο για το 334. Πέρας. 28 υπέρ 29 κατά απορρίπτεται. Απορρίφθηκε. 335 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 329. Έλεγχο το δεύτερο τμήμα. Παρακαλώ. Δεύτερο τμήμα. 325. 335 μάλλον. Πέρα τη ψηφοφορίας, 33, 33 υπέρ 24 κατά εγκρίνεται. 329 υπέρ κατά Αποχές. Κάποιες φορές ε, σηκώνονται λίγα χέρια. Ας ελέγξουμε λοιπόν. 326. Όχι, 329. Με συγχωρείτε. 329. Έλεγχο. Πέρας. 33 υπέρ, 25 κατά εγκρίθηκε. Περνάμε απευθεία στη συμβαστική 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 369 υπέρ. Ο κύριος Μπουτικόφερ. Συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε. Ψηφίσατε το 326. Κάνατε την ψηφορία. Κοιτάξτε, καταπίπτει γιατί 330 και 331 εγκρίθηκαν. Εξού και καταπίπτει. Εφόσον αυτές οι δύο εγκρίθηκαν, ε, καταπίπτει. Περνάμε στην 369. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 359. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 343. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 363. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 364 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 374 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 370 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 373 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 375 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 376 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχο για το 376. Πέρας της ψηφοφορίας 376-22 προς 32 απορρίπτεται. 383 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 392 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 395 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 300 έλεγχο για την 395. Άρχεται η ψηφοφορία, παρακαλώ. Πέρας. 32 υπέρ, 24 κατά, εγκρίνεται. Επειδή είναι κάπως μακροσκελής η ψηφοφορία σας, παρακαλώ βοηθήστε με, υψώνοντας τα χέρια σας γιατί αλλιώς 396, 396 υπέρ, κατά, έλεγχος. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά πρέπει να επαληθεύσουμε. Πέρας. 21 υπέρ, 36 κατά, απορρίπτεται. 397 υπέρ κατά απορρίπτεται. Έλεγχο, έλεγχο για την 397. «29, 29 απορρίπτεται». Τι να κάνουμε. 25 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 408 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 409 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 220 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 220. Πέρας. 24 υπέρ 31 κατά απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την 417 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 420 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 426 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 427 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Έλεγχος για την 427 παρακαλώ. Πέρας. 30 υπέρ, 25 κατά, εγκρίνεται. 427. 430 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 432 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία 499. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, 502. 502 υπέρ, 502. 502-502. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Κιούζα. Πέρας. 24 προς 31 απορρίπτεται. Μπέλετ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 479 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 481 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος για την 481 για να είμαστε βέβαιοι για τις πλειοψηφίες. Πέρας. 23 υπέρ, 31 κατά. Απορρίπτεται. Και τώρα ένα σύνολο. 482, 483, 484, 485. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 503 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μοιάζει να εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να ελέγξουμε. Πέρας. 23 υπέρ, 32 κατά, απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 26 και 24 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές έλεγχος έλεγχος για την 27. Κιούζα. Πέρας. 31 προς 26 εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, δεν είδα τίποτα. Να ελέγξουμε για την 32. Πέρας. 29, 29. Απορρίπτεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές δεν βλέπω. Οπότε κάνουμε έλεγχο για την 42. Πέρας. 27 προς 29. Απορρίπτεται. 44. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 49. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 έλεγχος. Πέρας. 28 υπέρ, 29 κατά, απορρίπτεται. 53, 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58. Τι θέλετε, έλεγχο για τον 60? Έλεγχο. Πέρας. 24-34 απορρίπτεται, με συγχωρείτε, απορρίπτεται η 60-58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έλεγχο για την 58, παρακαλώ. Πέρας. 26 προς 30 απορρίπτεται η 28, η 58 συγγνώμη. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. τα 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. τα 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ένβη 22. Ένβη 22. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ένβι 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 11 υπέρ κατά αποχές. Ρέτζι 11 άρχεται η ψηφοφορία. Κιούζα. Πέρας. 31 υπέρ 24 κατά εγκρίνεται. Ρέτζι 11. Ρέτζι 20 υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος για τη Ρέτζι 20. Γιατί κάποιοι μετακινούνται. Πέρας. 26 υπέρ 30 κατά απορρίπτεται. Ρέτζι 24 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Άγκρι 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 20 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος. Έλεγχος για την Άγκρη 20. Κιούζα. Πέρας. 29 υπέρ, 26 κατά, εγκρίνεται. Άγκρη 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική, άρχεται ψηφοφορία. 49 υπέρ 7 κατά, μία αποχή, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ωραία. Ωραία. Και τώρα έκθεση Τσίτσεστερ. Έκθεση Τσίτσεστερ. Δύο λεπτάκια. Να πιω λίγο νεράκι. Pronti per il voto? Rapporto Chichester, bene. Compromesso 1. Έκθεση Chichester, λοιπόν. Ε, η συμπτωπολογία 1, συμβαστική 1, υπέρ, κατά, Αποχέ, εγκρίνεται. Πρώτη τροπολογία, υπέρ, κατά, Αποχέ, εγκρίνεται. 2, υπέρ, κατά, Αποχέ, εγκρίνεται. 65, σε δύο τμήματα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 87 89 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 86 και 90 μαζί. 86 και 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα είναι πολλέ οι σελίδε. Φτάνουμε στην 116 και 16 μαζί. 116 και 16 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21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 Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39 και 40 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Όχι, φτάνει. Τέσσερα. Δεύτερο τμήμα δεν χρειάζεται να ψηφιστεί. Τέσσερα. Budget υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σαράντα τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές Ε, δεν είδα να σηκώνονται χέρια για τη 44. Άρχεται η ψηφοφορία. 44. Πέρας. 15-38 απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56, 7, 57, όχι, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ Α, ξέχασα την 8. Πρέπει να ψηφίσουμε και την 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, ας ξαναψηφίσουμε, 63 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέλος ε, της προφορίας, ηλεκτρονική ψηφοφορία τελική, άρχεται, πέρας. Πέρας. 51 υπέρ, Καμία αρνητική ψήφο, έξι αποχέ εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Περνάμε στο επόμενο σημείο με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ωραία. Πέρας. Εγώ Έβγαλα την κάρτα μου. Ένα σελ και Παραπάνω ένα είναι στο ΕΛΚ. Ωραία. Πέρας. 52 υπέρ, 0 ψήφι κατά. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ωραία. Περνάμε στην ψηφοφορία της Μισελ Ριβαζή. Παρακαλώ να ξεκινήσουμε με τις πρώτες δύο ψηφοφορίες, 8 και 9. Όλοι έτοιμοι για τη Ριβάζη. Ωραιότατα. 8 και 9 μαζί. Περ. Κατά. Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 55. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 56. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 57. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 58 και 59 μαζί. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 60 υπέρ κατά απορρίπτεται 61 υπέρ κατά απορρίπτεται 63 και 86 μαζί υπέρ κατά απορρίπτονται 62 υπέρ κατά απορρίπτεται 12 υπέρ κατά εγκρίνεται 11 υπέρ κατά εγκρίνεται 65 υπέρ κατά εγκρίνεται 66 υπέρ κατά εγκρίνεται 67 υπέρ κατά εγκρίνεται 13 όχι 68 υπέρ κατά εγκρίνεται 14 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβαστική υπαριθμών 2. Υπέρ κατά εγκρίνεται. 72. Υπέρ κατά απορρίπτεται. 17 και 73 μαζί. Υπέρ κατά απορρίπτονται. 74. Υπέρ κατά απορρίπτεται. 75. Υπέρ Κατά. Απορρίπτεται. 77. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 76. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 78. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται ηλεκτρονικός έλεγχος για τη συμβαστική υπαριθμών 3. Ψηφίζουμε. Πέρας. 21, 33 απορρίπτεται. 81. Α, α, συμπαθάτε με. Πάμε στο 79. απορρίφθηκε η συμβαστική τριά Και γι' αυτό και θα ψηφίσουμε 79 και 80, 79. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. αποχέ, εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. απόχέ, απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε την 88. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 89. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 90. Υπέρ, κατά, αποχές. Θα γίνει ηλεκτρικός έλεγχος για το 90. λάθος ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Χώρα ούνα. Allora, eh, Πέρας. 27, 30. Απορρίπτεται. 91. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές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 Απορρίπτεται. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Όχι, όχι, όχι, εγκρίνεται, διορθώνει ο πρόεδρος. Και θα κάνουμε έλεγχο για το 99. Votazione chiusa. Πέρας. Α, απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 26 100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 102. Υπέρ, κατά. Αποχές μας για το 102. Πέρας. Η 27-30 απορρίπτεται. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 104. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 105. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 107 εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και τον έλεγχος για ποιο? 113. Θέλει η εισηγήτρια. Ψηφίζουμε. ένας παραπάνω από το ΕΛΚΑ. 28-26 εγκρίνεται. Το 3 Το 114 το ψηφίσαμε και πάμε στο 21. Υπέρ. 115 υπέρ κατά αποχές Για να κάνουμε το για όσον αφορά το 115. votazione. 15 πέρασε τη ψηφοφορία. Η 28-27 εγκρίνεται. Il 116. 117 υπέρ. Κατά. Αποχές. 117 ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρας. 33-23 εγκρίνεται. 117 και τώρα θα ψηφίσουμε από κοινό 117, 118, 119 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 120 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για το 120. 48 48-9 εγκρίνεται από κοινού. 121 και 122 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και τον 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 127 23 ήταν πριν. όχι 123. Απορρίπτεται το 127. Και 128 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για τη συμβαστική 5. Check sul compromesso 5. Votazione chiusa. Πέρα τη ψηφορία. 22, 33. Μπορείτε και τώρα. Πάμε. Στην τροπολογία 131. Συγγνώμη, 141. Υπέρ. Κατά. 141. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Χιούζα. Πέρας. 27, 28. Απορρίπτεται. Κατόν σαράντα έξι. Υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 28. Συγητής. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 142 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Για τη συμβαστική 7 θα κάνουμε έλεγχο, ψηφίζουμε. Πέρας ή 29, 27. Εγκρίνεται. Εγκρίθηκε η 7 και πάμε επομένω. 153 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Α, απορρίπτεται. Αλλά για τα 153 θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ψηφίζουμε. Πέρας 31-26. Εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωται. 156 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36 ε, εγκρίνεται, 37 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 38 Μου λέει ότι ξέχασα, παρέλειψα μία ε, τροπολογία, την 157. Την ψηφίζουμε αυτήν που ξέχασα. Την βρήκατε. Υπέρ. 157. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και τώρα από κοινό την 38, 39, 40 και 41. Όλες μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Εγκρίνεται μάλλον. 160, α, όχι, όχι, όχι. 161 λέει ο 161. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται έλεγχος για το 166. Πέρας. 27-28 απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μαζί η 1 και 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Απορρίπτονται μάλλον. Δεν θα ψηφίσουν τη 43 γιατί ήδη έχει καλυφθεί. Και πάμε τώρα στην 3. 4. Υπέρ κατά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 Τελική ψηφοφορία. Ναι, έχετε το λόγο. Ναι, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι το όνομά μου δεν περιλαμβάνει. Πριν τελική ψηφοφορία, συνάδελφοι, θέλω κάτι να πω στην πρώτη, ότι το όνομά μου δεν αναφέρεται στο κείμενο. Ναι, καλά θα τη λάβουμε υπόψη και ως πρόεδρος θα το φροντίσω. Και τώρα πάμε στην τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. 32-23. Μία εποχή εγκρίνεται. Καλώς και τώρα προχωρούμε. Έχουμε και άλλες σοβαρίες. Έχουμε ακόμα κάτι δουλίτσες για το πρωί. Περνάμε στην έκθεση Φιώνα Χολ. Εάν είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε αμέσως. Έτοιμοι όλοι. Ωραία. Τέλεια. 42. Παρακαλώ. Πρόεδρε, εξώ αν κατάλαβα από αυτά που μας είπε η γραμματεία, οι συμβαστικέ θα ψηφιστούν πρώτε. Ιδάλω θα ψηφίσουμε πράγματα τα οποία θα καταπέσουν ε, αν εγκριθούν οι συμβιβαστικέ προτάσει. Και η γραμματεία μου είπε ότι αυτό επρόκειτο να κάνουμε παρά τον κατάλογο ψηφοφορία και τη σειρά που αναφέρονται οι τροπολογίε, πρώτα πρέπει να ψηφίσουμε τι συμβιβαστικέ. Να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό μου είπε η γραμματεία, όντως. Δεν το γνώριζα το θέμα, τώρα το συζήτησα με τη γραμματεία. Για να μην υπάρξει προηγούμενο. Εάν συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι, θα συμφωνήσουμε πρώτη-πρώτη την συμβαστική εννέα Και μετά τα υπόλοιπα. από την 1 ως την 9, εάν συμφωνείτε όλοι οι συνάδελφοι, εάν οι συμβιβαστικές και να αλλάξουμε τον κατάλογο των ψηφοφοριών, πρέπει να ξεκινήσουμε με τις συμβαστικές 1 έως 9 και μετά ψηφίσουμε τις υπόλοιπες τροπολογίες. Εάν συμφωνείτε όλοι με αυτό, διότι είναι κάτι το καινούργιο. Ψηφίζουμε τι συμβαστικέ από την 1 ω την 9 και μετά βλέπουμε τι έχει καταπέσει και ψηφίζουμε τα υπόλοιπα. Συμφωνείτε, καμία αντίρρηση. Ωραία. Εφόσον όλοι συμφωνείτε, ξεκινάμε με τη συμβαστική 1, υπαριθμόν 1. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 3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 devait être beaucoup attentif de moi donner la juste liste de vote après. Bene, perfetto. Allora, bene, partiamo con il voto. Emendamento... Ξεκινάμε την ψηφοφορία. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 και 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45, 47 συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 7, 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την 7. Check 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πάλι ένας από το ΕΛΚ είναι υπεράριθμος. «22 υπέρ, 34 κατά, απορρίπτεται». «44 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται». 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος, έλεγχος για την 51. Παρακαλώ. Πέρας. 29 υπέρ, 28 κατά, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Περνάμε στην 73 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για την 73. Πέρας. 30 υπέρ 24 κατά. Εγκρίνεται. ...79 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχο για την 96. Πέρας. 30 υπέρ 26 κατά εγκρίνεται. Εκατόν δέκα. Εκατόν δέκα. Μισό λεπτό. Ναι. Εκατόν δέκα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατόν έντεκα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100, συγγνώμη, 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Έλεγχος για την πρώτη τροπολογία. Πέρας. 26 υπέρ 31 κατά. απορρίπεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 29 Πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίν, απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Okay. Πέρας. Voilà. Πέρας. 51 υπέρ, 5 κατά. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Bene. Ωραία. Ψηφίζουμε τώρα Πίπερ. Ετοιμαζόμαστε. Tutti pronti, relazione Piper. Όλοι έτοιμοι για την έκθεση Πίπερ. Compromis Είναι tutti pronti? Prego, Mr. Johnson. Παρακαλώ, ο κύριος Τζόνσον. Έχω ένα αίτημα, η τροπολογία 21 να ψηφιστεί σε τμήματα, γιατί η συμβιβαστική 1 αναφέρεται στους στόχους του 2025 και εγώ αναφέρομαι στους στόχους του 2020. Άρα πιστεύω ότι θα πρέπει να ψηφιστεί ξεχωριστά η τροπολογία 21. Αυτό ζητάω. Πίπερ, Παρακαλώ, κύριε Πίπερ. Λέμε στη συμβαστική ότι επιβεβαιώνουμε το στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020, το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και δεν θέλουμε άλλη αλλαγή μέχρι το 2020, αλλά δεν έχουμε συγκεκριμενοποιήσει τα πράγματα. Δηλαδή, εξακολουθεί να ισχύει ο στόχος για τα γραμμάρια και άρα αν ισχύσει η συμβιβαστική πρόταση και περάσει, δεν θα ισχύει πλέον αυτή η τροπολογία. Δεν θα μπορούμε να την ψηφίσουμε. Αυτό επιβάλλει λογική. Allora, in base ai documenti preparati... Βάσει των εγγράφων που μου έχει ετοιμάσει και η γραμματεία, ε, βρίσκομαι ενώπιον τη εξή κατάσταση. Αν ψηφίσουμε την πρώτη συμβαστική και εγκριθεί, οι υπόλοιπε τροπολογίε 22, 21 κλπ. κλπ. θα κατέπιπτο, κατέπιπταν μέχρι την 30 Αυτά μου λένε τα στοιχεία που με έχουν ετοιμάσει. Το ίδιο λέει και ο εισηγητή. Οπότε, ω συνήθω, ο κανόνα που ισχύει είναι ότι εάν κάποιο συνάδελφο θεωρεί ότι αυτό δεν καλύπτεται, και βάσει των ενδείξεων της γραμματείας είπαμε τροπολογίες από την 1 έως την 29 και αυτή συμπεριλαμβανομένες καλύπτονται από την ε, συμβεβαστική. Ο κύριος Τούρμερ. Νομίζω ότι φαίνεται ότι υπάρχουν δύο καταλεκτικές ημερομηνίε, δύο προθεσμίες. Ίσως να τις ψηφίσουμε και τις δύο. Αν περάσει, πέρασε. Αν δεν περάσει, δεν πέρασε. Intanto την πρώτη τροπολογία λοιπόν, συμβαστική 1. Και να δούμε τι θα γίνει. Συμβαστική 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κατ' εμέ όλες οι υπόλοιπες τροπολογίες καταπίπτουν. Υπήρξε ένα συγκεκριμένο αίτημα βέβαια το οποίο μπορούμε να το ψηφίσουμε. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώ. Αυτό είναι ο κανονισμό. Εάν υπάρχει αίτημα, μπορεί να ψηφίσει, μπορούν να ψηφίσουν οι παρόντε, αλλά κατά κατεμέ όλε έχουν καταπέσει. Δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα, οπότε περνάμε στην 30. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 33. Υπέρ. Όχι, όχι, με συγχωρείτε. 31. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 37, 37 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την 5. Votazione chiusa. Πέρας. 40 υπέρ, 14 κατά, εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά 2-2 του εισηγητού υπέρ κατά εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική. Παρακαλώ. Bene. Ωραία. Τελική ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντε. Τέλεια, τέλεια. Πέρα τη ψηφοφορία. 36 υπέρ 12 κατά. Μία εποχή εγκρίνεται συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ωραία λοιπόν, ολοκληρώσαμε με τις πληροφορίες, πέντε λεπτά για να, διά, για διάσει αίθουσα και μετά έχουμε την έκθεση Τσίτσεστερ. Όποιος θέλει να φύγει, να φύγει αμέσως. Bene. Purtroppo... Ωραία. Δυστυχώς... Το θέμα είναι ότι όσοι έρχονται να παρακολουθήσουν τις προφορίες καθυστερούν να βγουν από την αίθουσα. Τέλος πάντων. Ξεκινούμε αμέσως. Ζητώ όλοι να σοπάσετε. Να ακούσουμε τον συνάδελφο Τσίτσεστερ, εισηγητή για την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη. Μια βιοοικονομία για την Ευρώπη. Παρακαλώ. Κύριε Τσίτσεστερ, έχουμε μισή ώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχετε το λόγο. Well, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περιμένω να βγουν όλοι από την αίθουσα και να μιλήσω μετά πιο διακριτικά. Να ευχαριστήσω τους λίγους και εκλεκτούς που έμειναν. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση για μια έκθεση της ε, Επιτροπής Περιβάλλοντος και θα πρέπει να πω ότι η πρώτη μου σκέψη είναι να αμφισβητήσω το τι έχει να κάνει η Επιτροπή Περιβάλλοντος με οποιαδήποτε οικονομία. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, πρόκειται για την βιοοικονομία. Έως ε, εκ τούτου προσπάθησα να καταρτήσω μια γνωμοδότηση από την πλευρά προφανώς της Επιτροπής Βιομηχανίας και να αναφέρω κάποιους τομείς όπου πιστεύω ότι μπορούμε να συμβάλλουμε με χρήσιμο τρόπο στη συνολική έκθεση, εντοπίζοντας τομείς στους οποίους η βιοοικονομία θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την εσωτερική αγορά, για την οικονομία, για την ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, για την αγορά εργασίας. Ε, νομίζω ότι αυτά είναι όροι με τους οποίους δεν ε, είναι απόλυτα εξοικειωμένη η Επιτροπή περιβάλλοντο. στο, στην αιτηλογική σκέψη την πρώτη αναφέρω τα πιο σημαντικά θέματα, όπου υποθυμίζω ότι είναι σημαντική η οικονομία στα πλαίσια της ιστορικής αγοράς που συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα, τη μείωση της εξάρτηση από τα, από τις πρώτες από την εισαγόμενη ενέργεια. Αυτό θεωρώ είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερο σημείο που τονίζω είναι στο σημείο 6, παραγραφός 6, ότι καλούμε την βιομηχανία να διαδραματίσει το ρόλο που της αναλογεί, την βιολογική ε, βιομηχανία, αναπτύσσοντας την, βιολογική, την βιοοικονομία. Γιατί χωρίς την καινοτομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν θα υπήρχε ιδιαίτερη πρόοδος. Πέραν τούτων, θεωρώ ότι όλα είναι αρκετά σαφή και προτείνω να την υπερψηφίσει η Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, συνάδελφε Τσίτσεστερ. Και τώρα το λόγο έχει ο συνάδελφο πρώτη Ο συνάδελφο Πρόντι. Ναι, ναι, ναι. Έχετε το λόγο, συνάδελφε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το έγγραφο και η έκθεση, διότι ο κλάδος της βιοοικονομίας έχει προοπτικές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Ακριβώς γιατί έτσι την είναι τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε την βιομάζα. Ως βάση για μια νέα χημεία, ούτως ώστε θα μπορούσαμε να υποκαταστήσουμε την πετροχημία, την πετροχημική το μητροχημικό κλάδο τέλο πάντων. Οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις δυνατότητες ούτως ώστε να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες. Και βεβαίως πρόκειται περί δηλώσεως αρχής ότι η προτεραιότητα στην χρήση του εδάφους θα πρέπει να παραχωρηθεί στην παραγωγή τέτοιων ουσιών, τέτοιων θρεπτικών ε, ειδών διατροφής, διατροφών, ούτως ώστε η χρήση του εδάφους για άλλους σκοπούς να διέπεται από, την, από τον έλεγχο της συμβατότητας. Αν δεν μεριά πάρα πολλά είδη βιομάζας ακόμα και στα πλαίσια της δασοπονίας που παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μέχρι σήμερα δεν έχουν ε, αναπτυχθεί. Οπωσδήποτε από πλευράς βιομηχανίας, από πλευράς της δικής μας επιτροπής ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι θα γίνει με την περισυλλογή, ε, με την ε, επεξεργασία αυτών των ουσιών που σχετίζονται με τα δάση. Οπότε μιλούμε τώρα για άλλη διαφορετική κατηγορία βιομάζας. Γιατί υπάρχουν ε, κάποια εδάφη τα οποία έχουν υποστημόλυνση και εκεί δεν μπορούμε να έχουμε Καλλιέργειε που αποσκοπούν στη διατροφή. Θα πρέπει επομένω να περάσουν αυτές τι περιοχέ από, από έναν καθαρισμό, μια κάθαρση τέλο πάντων ε, ριζική και βαθμία και έτσι αυτό να γίνει με καλλιέργειε που συμβάλλουν στην παραγωγή ενέργειας. Όλα θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα γιατί ακριβώς πρόκειται για μεγάλε εκτάσει που έχουν υποστεί αυτή την μόλυνση και άρα μπορούν τώρα να βοηθήσουν την βιοοικονομία. Οπότε, να καταλήξουν τελικά και για εκμετάλλευση που να αποσκοπεί στην παραγωγή των διατροφής για τον άνθρωπο. Βεβαίω, πρόκειται για καινοτομίες σημαντικές για αυτά τα κέντρα της ε, in sostituzione eh, della petrolchimica. τις εγκαταστάσεις της πετροχημικές για ε, τα, τα βιοδηληστήρια. Ούτω ώστε βλέπουμε ότι πρέπει έχουν, υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικέ προοπτικέ. και έχει μέλλον λοιπόν στο θέμα. Ευχαριστούμε κύριε, κύριε Πρόντι ο συνάδελφος Κράμερ, ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, νομίζω ότι ο εισηγητής και μας υποβάλλει μία πρόταση η οποία θεωρώ ότι είναι σωστή και κατάλληλη για το ζήτημα αυτό. Η βιοοικονομία ασφαλώς και θεωρώ ότι προσφέρει ευκαιρίες τις οποίες θα πρέπει να δράξουμε, αλλά δεν θα ήθελα να υπερφορτώσουμε, αν θέλετε, την Ευρώπη με μια νέα στρατηγική. Να σας υπενθυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δραμολογήσει πάρα πολλές καινούργιε στρατηγικές, οι οποίες έχουν προκαλέσει και ανάγκη προσαρμογής της νομοθεσίας. Για παράδειγμα, για τα βιοκαύσιμα, η σχετική στρατηγική χρειάστηκαν πάρα πολλές αλλαγές μέχρι να καταλάβουμε ότι δημιουργούμε ουσιαστικά έναν ε, ουσιαστικά αντιδεοντολογικό ανταγωνισμό για τις αγροτικές πρωτεσίλες ε, μεταξύ δηλαδή των καυσίμων και των ε, τροφίμων. όλα αυτά χρειάστηκε να τα προσαρμόσουμε σε ό,τι αφορά τη βιομάζα, σε ό,τι αφορά, αφορά τις εκπομπές, γιατί δεν μπορούσαν να εκπληρώσουν αυτά που είχαμε υποσχεθεί. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα αυτό στις πραγματικές του διαστάσεις, ως μία δυνατότητα να επιλέξουμε κάποια πραγματικά προβλήματα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι τομείς εφαρμογή όπου διαπιστώνουμε ότι η αντικατάσταση των ορεικτών καυσίμων ε, είναι δυνατή από βιολογικά, από βιο καύσιμα. Δεν ξέρω όμως σε τι βαθμό μπορεί να γίνει αυτό. Θα έπρεπε, θεωρώ, να κοιτάξουμε πιο πολύ θέματα έρευνα και να προσέξουμε γιατί μπορεί με τις πολλαπλές στρατηγικές που επιβάλλουμε να ε, αναιρέσουμε την ε, οικονομία της αγοράς. Είμαι σχετικά βέβαιος ότι θα είναι αρκετά ξεκαθαρισμένη αν θέλετε η άποψη και η τοποθέτηση της επιτροπή Περιβάλλοντος και γι' αυτό πιστεύω ότι εμείς ως Επιτροπή Βιομηχανία θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να καταλάβουμε ότι είναι μια ευκαιρία, αλλά δεν πρόκειται για ένα μαγικό όπλο. Υποστηρίζουμε λοιπόν αυτά που προτείνει ο εισηγητή, ενδεχομένω να υπάρξει ανάγκη να, να καταθέσουμε κάποιε προπολογίες, αλλά θεωρούμε ότι το έγγραφο στη μορφή που έχει σήμερα είναι επί της ουσίας επαρκές. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να παρέμβει, λέει η Grazie, signor Presidente, onorevoli, buongiorno. Καλημέρα σας αγαπητοί. Πολύ χαίρομαι που ήρθα εδώ να σας ακούσω και επίσης να σας πω ποια είναι η δική μας συμβολή για την ελλογοστρατηγική. Να σας πω πρώτα πρώτα ότι η βιοοικονομία δεν είναι αυτόνομος τομέας. Είναι κάτι το οποίο καλύπτει άλλους κλάδους της οικονομίας, ε, την ε, διατροφική βιομηχανία, την ε, γεωργία, την αλληλεία. διάφορους δηλαδή κλάδους οι οποίοι χρησιμοποιούν τους φυσικούς πόρους. Και αυτό το σύστημα το οποίο τώρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ερώτημα είναι ότι να δούμε πώς θα μπορέσουμε ως στόχο να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και ταυτοχρόνως να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια βιωσιμότητα μακρόπνοη. Οπότε αυτό εδώ έχει τονιστεί επανελειμμένα. Και επίσης είναι σημαντικό να προσέξουμε αυτούς τους κλάδους αυτή την, οπτική γωνία, δηλαδή πώς θα έχουμε τεχνολογική ανάπτυξη, οπότε θα πρέπει να προσέξουμε το πόσο είναι δύσκολο να, ε, να, να που αφορούν τα ιδιατροφής και τους άλλους. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα προωθήσουμε την τεχνολογία την λεγόμενη δευτέρας ή και τρίτης γενεάς. Ε, αυτό το οποίο ακριβώς ανέφερε και ο κύριος Πρόντι σε σχέση με το πώς θα μπορέσουμε να άρουμε αυτή την αντίθεση μεταξύ των, δύο δραστηριοτήτων, των δύο ειδών δραστηριοτήτων για ιδιατροφής και όχι. Και επίσης θα πρέπει από πλευράς καινοτομία να προσέξουμε και άλλες μεθόδους, άλλους τρόπους ε, παραγωγής, δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει με την πράσινη χημεία και στη συνέχεια να μπορέσουμε να έχουμε αυτό το, το, το φαινόμενο της σόρευσης των ε, στόχων και επιτυχιών και ε, να δούμε τι γίνεται από πλευράς ε, εθνικού επίπεδου για αυτές τις στρατηγικές που αναπτύσσονται σε κρατημέλη, σε περιφέρειες ούτω ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αυτό το οποίο ονομάζουμε smart specialization. ακριβώ για κάποιε περιφέρειε που θέλουν να εκμεταλλευτούν καλύτερα του φυσικού πόρου. Και τώρα στον Όρφο για να κάνει τα κρατικά σχόλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και του συναδέλφου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι ε, παρεμβάσει του. για την ε, βιομηχανία πετροχημικών. Θα ήθελα να σχολιάσω γιατί ο γεωλόγος μέσα μου διατείνεται ότι το πετρέλαιο και ο άνθρακας και το αέριο αρχικά ήταν τμήματα της βιοσφαίρας που στη συνέχεια μετατράπησαν στα καύσιμα τα οποία σήμερα χρησιμοποιούμε. Σύμφωνα όμως με τον κύριο Πρόντι ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το τι γίνεται και πέρα από τα ορεκτά καύσιμα και την χημική βιομηχανία και να αναπτύξουμε νέες τεχνολογίες χρησιμοποιώντας βιώσιμα συστήματα παραγωγής. Και έτσι περνάω στο δεύτερο σημείο. Για την ανάγκη να γίνει διάκριση μεταξύ της παραγωγής τροφίμων και την χρήση γεών για άλλες μορφές βιοοικονομικής δραστηριότητα, βιομάζα και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται λίγο κοινή λογική. Θα πρέπει να εξετάσουμε τη χρήση γης και να δούμε όταν δεν χρησιμοποιείται η γη για παραγωγή τροφίμων, μήπως θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλη, για άλλα είδη παραγωγής. Αυτό μου φαίνεται αρκετά εύλογο. Ελπίζω να μην αντιμετωπίσουμε δυσκολίε σε ό,τι αφορά άλλες νομοθεσίε για τον ορισμό της χρήση των γεών. Να σας ευχαριστήσω συνάδελφοι, αν έχετε οποιαδήποτε προσθήκη να κάνετε. Βεβαίω ε, προσβλέπω στις ε, τροπολογίες σας να ευχαριστήσω τον κύριο Κράμερ για τα καλά του λόγια και ευχαριστώ και την Επιτροπή που ορίζει το πλαίσιο της πρότασης. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε για την δημιουργία ευημερία, τη δημιουργία θέσεων εργασία, τη δημιουργία νέων τεχνολογιών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Τσίσαστερ. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 25 Μαρτίου την Μεσημβρία. Και τώρα. Επίσης να σας ενημερώσω σε όσους μείνατε εδώ ότι κατά την συνάντηση των συντονιστών αποφασίσαμε να κάνουμε μία μίνι ακρόαση αφορά τις ε, βιομηχανικές στρατηγικές ούτως ώστε να αξιοποιηθούν όλες οι δραστηριότητες που καλύπτονται από τον Γαλιλαίο. Θα γίνει αυτό προσεχώς. Επίσης είπαμε ότι έχουμε κάποια αλλαγή ε, την 17η δεκάτου δεν θα κάνουμε συνεδρίαση αλλά θα κάνουμε στις 14 αντί 17, 14 επίσης αποφασίσαμε να αναλυθεί μία μελέτη ε, για τη δουλειά της ε, ΕΝΒΗ για την e-society, ηλεκτρονική κοινωνία και θα έχουμε επομένω ε, συνεργασία με την Ιντερ. Επίσης, έχουμε αναθέσει δύο, ε, δύο, δύο εκθέσεις για το GNSS και επίσης θα πρέπει να ανατεθεί μια έκθεση για τη δέσμη τηλεπιονιών και επίσης και για την ε, ψηφιακή πολιτική και επίσης όσον αφορά την ε, βιομηχανία σχέση με το διάστημα και τέλος εγκρίναμε μια γνωμοδότηση σε σχέση με την ασφάλεια των προϊόντων. Αυτά. Και στις 3.30 θα τα πούμε με την Επιτροπή Κρούς. Στις 3.30. 3.30. Καλή όρεξη.